τα πιστοτικά ιδρύματα. Αν έχουμε τέσσερα ε, μέλη, αν, αλλά μιλάμε με μια φωνή, ε, τότε καλύτερα θα ήταν να έχουμε έτσι, πιο ενιαία φωνή παρά διαφωνίες. Ναι, αν θέλουμε να παίξουμε το ρόλο μας σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, πρέπει φυσικά να έχουμε ενιαία θέση, να μιλάμε με μια φωνή. Σιλβί, θες να πεις κάτι άλλο, έχεις ακόμα ένα λεπτό. Από την Ευχαριστώ. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις. Πρώτον, για το ERS, η FRS 27. Υπήρχαν κάποια προβλήματα που έπαιξαν ένα ρόλο πώς χρησιμοποιούνται, πώς χρηματοδοτούνται συγγνώμη, οι εταιρείε ειδικού σκοπού. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η δική σας προοπτική ως επικεφαλής του ΕΦΡΑΓ για τα θέματα αυτά, πώς θα τα αντιμετωπίσετε και σε σχέση με αυτό μια γενική ερώτηση για τα λογιστικά πρότυπα όπως είπατε και εσείς υπάρχουν αυτοί οι κύκλοι boom and bust, οι οποίοι μπορούν να παίξουν προκυκλικό ρόλο. Δηλαδή, εάν κάποια στοιχεία χρησιμοποιούνται ως εγγυήσει ε, για τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων, τότε μπορεί να συμβάλλουν σε αυτές τις φούσκες. Πώς θα θέλατε να το αντιμετωπίσετε. Γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε απλώς μία φιλοσοφία περισσότερο απλώς να εγγράφουμε τα στοιχεία σε ένα κατάλογο. Και οι οργανώσει μέλη του ΕΦΡΑΓ και ε, οι ομάδες εργασίας αποτελούνται κυρίως από εμπειρογνώμονες που προέρχονται από τις οργανώσεις παροχής συμβούλων Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτές τις ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων. Για την πρώτη σας ερώτηση. Για τις εταιρείες ειδικού σκοπού. Πάντα θεωρούσα ότι είναι λάθος να λειτουργούν εκτός ισολογισμών. Αυτή είναι σοβαρή παραβίαση της πιστής εικόνας, της εικόνας του true and fair. Αν θέλουν οι ισολογισμοί να δίνουν μια σωστή εικόνα της λειτουργίας των επιχειρήσεων για να το ξέρουν όλοι οι επενδυτές, οι μέτοχοι και τα λοιπά, οι εργαζόμενοι, τότε πρέπει να τα λέμε ότι υπάρχει μια εταιρεία ειδικού σκοπού η οποία μπορεί να σημαίνει υψηλό κίνδυνο ενδεχομένω. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να γίνει. Γιατί στο παρελθόν ήταν πολύ σοβαρό θέμα, τώρα πια δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Και στη Γερμανία το είχαμε αυτό. Και εδώ δεν ε, είχαμε αποτυχία μόνο των προτύπων, αλλά και των υποπτικών φορέων. Θα έπρεπε και αυτοί να το έχουν λίγη υπόψη. Δεν είναι δυνατό να λέμε για κάποια γερμανική εταιρεία με μια υποσημείωση, με ένα αστερίσκο υπάρχει μια ειδική εταιρεία στην Ιρλανδία. Δεν είναι σωστό αυτό για τις τεχνικές ομάδες εμπειρογνωμόνων. Όπως λέει ε, και το όνομα αυτών των επιτροπών και ομάδων, πρέπει να είναι εμπειρογνώμονες αυτοί που συμμετέχουν. Δεν έχω συναντήσει ακόμη τα μέλη, αλλά απριόρι. Δεν θεωρώ ότι θα ήταν επιζήμιο, λαθασμένο, να συμμετέχουν λογιστές ή άλλοι εμπειρογνώμονες. Γιατί πρέπει πραγματικά να δώσουν ειδικευμένε συμβουλές η πρότασή σα για τη συμμετοχή της ε, κοινωνία των πολιτών, πώς θα μπορούσε να συμμετάσχει. Η κοινωνία των πολιτών θα μπορούσε να συμμετάσχει στο καθορισμό των στόχων. Τι θέλουμε να επιτύχουμε μέσω των προτύπων. Εκεί θα πρέπει να συμμετάσχει, να μας βοηθήσει να ορίσουμε το ευρωπαϊκό κοινό καλό και πώς θα πρέπει να αποτυπωθεί στα πρότυπα. Δεν νομίζω ότι έχει έννοια να βάλουμε 10 μέλη των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Πρέπει να είναι εμπειρογνώμονε. Δεν είναι δυνατόν να του αντικαταστήσουμε με απλώ εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών. Εκτό φυσικά αν είναι και εκείνοι εμπειρογνώμονε. Βεβαίω. Πάνω τότε δεν θα τίθε το θέμα. Δεν θα τίθε το θέμα, θα ήταν εμπειρογνώμονε που αντικαθιστούν άλλου εμπειρογνώμονε. Πρόεδρο. Α, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είπατε ότι το πρόβλημα με τη διάταξη ERS 27 κάπως καταργήθηκε. Μπορείτε να εξηγήσετε λίγο περισσότερο. Απάντηση Κρίντς. Από όσα γνωρίζω, δεν είναι πια δυνατόν να παραμένουν αυτές οι εταιρείες ειδικού σκοπού εκτός ισολογισμών και να μην, ενδιαφε... και να μην αναφέρονται μέσα στον ισολογισμό δηλαδή της εταιρείας. Sven των πράσινων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, πρώτα εκφράζω τη χαρά μου για την υποψηφιότητά σου, η οποία υποψηφιότητα νομίζω ότι είναι και δείγμα της κοινή μας επιτυχίας. Τα τελευταία χρόνια φέραμε ξανά και ξανά το θέμα στην επικαιρότητα, μέχρι ότου μάλιστα να βάλουμε και στο αποθεματικό ένα μέρος του προϋπολογισμού της ΕΦΡΑΓ και το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβάλλει τώρα την δική σου υποψηφιότητα συναποτελεί δική μας επιτυχία. Ευχαριστώ λοιπόν την χαρά μου. Υπάρχει βέβαια και αυτή η ιδέα στην οικονομική επιστήμη των εξωτερικοτήτων και γι' αυτό παρακολουθούμε τώρα και την πολιτική σου οικογένεια, τους φιλελεύθερους δηλαδή, να έχουν εξωτερικεύσεις και σε άλλα κόμματα. Και εδώ έχω μια θετική εξωτερικότητα, στο πω έτσι. Πέρα από αυτό τώρα. Κέρια θέματα για τα πρότυπα είναι αυτά που τίθεται και βέβαια και της δημοκρατικής ευθύνης. Τώρα, η ΕΦΡΑΓ και ο IASB είναι παραδείγματα για το πώς η δημοκρατία υπάρχει ακόμα τα παγκοσμιοποιημένα θεσμικά όργανα. Θα ήθελα τώρα να μάθω πώς θα συμβάλλεις ώστε μέσα στα πλαίσια της ΕΦΡΑΓ να υπάρξει μια πολυφωνικότερη σύνθεση του οργανισμού. Βεβαίως σε ομάδα εμπειρογνωμόνων πρέπει να συμμετέχουν εμπειρογνώμονες. Δεν σημαίνει όμως ότι όλοι οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κλάδο της οικονομίας, διότι οι λογιστές δεν είναι Μάλλον διότι τα λογιστικά πρότυπα δεν είναι η ιδιοκτησία των επιχειρήσεων. Τα λογιστικά πρότυπα, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα είναι κυριότητας της ίδιας της κοινωνίας, γιατί εξυπηρετούν ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό θέλω να μου εξηγήσεις τώρα, αν θα το εξετάσεις από αυτή τη σκοπιά. Δεύτερο, η εκπροσώπηση σε διεθνές επίπεδο. Βεβαίως κατανοώ ότι σας ενοχλεί ότι η Κίνα δεν ορίζει με δημοκρατικό τρόπο τον εκπρόσωπό της που πηγαίνει στο IASB. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πως οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι δεν είναι δημοκρατικά εκλεγμένοι. Χρειαζόμαστε και εδώ λοιπόν μεγαλύτερη πολυφωνία, μεγαλύτερη δημοκρατική ευθύνη και θα ήθελα εκεί να ακούσω και τη φωνή της ΕΦΡΑΓ. Τέλος, διαρωτώ με, η ΕΦΡΑΓ το μέλλον θα τηρήσει αυστηρά τα όρια της εντολής της, να μην ανακατεύεται δηλαδή σε, άλλον, σε άλλες υποθέσεις. Όχι μόνο να επιβάλλει τα πρότυπά της σε άλλους φορείς, αλλά όπως το είδαμε και για τις χώρες, ότι η δηλαδή προβαίνει σε σχολιασμό, σε τομείς που δεν είναι διόλου υπόθεση δική της. Αυτά λοιπόν και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Απάντηση, απάντηση Wolf Ευχαριστώ πολύ βεβαίω για τις ευχές. Είπα και πριν ότι ακόμα δεν έχω δουλέψει ούτε μια ώρα στην ΕΦΡΑΓ. Εφόσον λοιπόν αναλάβω τα καθήκοντά μου εκεί, θα είναι νέο πεδίο αυτό δραστηριότητα για μένα. Η Technical Expert Group δεν ξέρω όποιο απαρτίζεται, πρέπει να το δω πρώτα. Και θα διαπιστώσω τότε δύο πράγματα. Πρώτο, η διαδικασία επιλογής των μελών είναι λογική, είναι σωστή, είναι διαφανής, είναι εύλογη. και το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής της επιλογής αρμόζει σε ένα οργανισμό τέτοιας ε, σημασίας. Τώρα, η εκπροσώπηση στον IASB. Κάθε χώρα που στέλνει εκπρόσωπο σε ένα τέτοιο συμβούλιο στο Λονδίνο θα κάνει βέβαια σύμφωνα με τα δικά της κριτήρια. Θα χρειαστεί να περιμένουμε αρκετά χρόνια νομίζω μέχρι ότου η Κινέζικη Δημοκρατία επιλέξει τους εκπροσώπους της με τον τρόπο που εμείς θεωρούμε δημοκρατικό. Όμως ακόμα τα μέλη στο ISP δεν διορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα, ναι, οι ίδιοι μάλιστα το επιλέγουν, λέει ο κ. Σκίγκολτ. Να φροντίσουμε τώρα να γίνει η υπόθεση αυτή πιο δημοκρατικά, πιο δημοκρατικά, τονίζω. Αυτό ναι, είναι κάτι που ευχαρίστως θα το εξετάσω και το σημειώνω το σχολείο σου. Όσον αφορά τώρα την ερμηνεία της εντολής της ΕΦΡΑΚ, εγώ δεν έχω καμία γνώση να έχει δηλαδή σχολιάσει η ΕΦΡΑΚ εκτός πλαισίων αρμοδιοτήτων της. Μεταξύ ΕΦΡΑΚ και Κοινοβουλίου θέλουμε να υπάρχει στο μέλλον ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων. Μπορώ να φανταστώ λοιπόν ότι ενδεχομένως θα φτάνουμε και σε κάποια όρια, δηλαδή θα φτάνουμε να σχολιάζουμε και κάποιες οριακές περιπτώσεις. Μπορεί ενδεχομένω να γίνει ε, δημοσιοποίηση μιας ε, γνωμοδότησης η οποία αγγίζει και κάποια όρια. Πρόεδρος Φέρβερ, ο κύριος Άνεμανς των μη εγγεγραμμένων. Δεν έχουμε ρηστικό μικρόφωνο. Ευχαριστώ. έχουμε πάρα πολύ την εμπειρία σας. Ήσασταν ευρωβουλευτής. Ξέρετε πάρα πολλά πράγματα και για τις επιχειρήσεις και για τα λογιστικά πρότυπα. Είσαστε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Νομίζω ότι ξέρετε το θέμα της γύρασης του πληθυσμού. Πρέπει να δουλεύουμε όλο και πιο πολύ μέχρι τα βαθιά γεράματα και είσαστε τέλειο παράδειγμα αυτού, αυτής της ανάγκης. Εντάξει, ίσως τώρα σας κάνω μία ερώτηση ως αδαής αλλά διερωτώ για τη χρησιμότητα αυτού του οργάνου. Πώς μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες ότι χρειάζεται τέτοιο όργανο όπως η Εφράγκα. Έχουμε ήδη τον Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Έχουμε το, το, έχουμε την Επιτροπή συμβουλευτικού χαρακτήρα για λογιστικά θέματα. Αναφερθήκατε στον κύριο Μαϊστάτ και στην ε, έκθεση του 2013. Η ΕΦΡΑΚ είναι παράρτημα του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, της ε, IASP. Στην έκθεση λέγεται ότι τα κριτήρια της IASB πάντα γίνονται σεβαστά από την ΕΦΡΑΓ. Κοιτάξτε, έχουμε άπειρα τεχνικά, τεχνικούς φορείς, ε, έχουμε τεχνικές ομάδες, έχουμε εποπτικές ομάδες. Τι σχέση έχει η ΕΦΡΑΓ με την IASB. Υπάρχει επικάλυψη. Πώς μπορώ να εξηγήσω τα πράγματα στους πολίτες. Ε, πώς μπορώ, πώς μπορώ να τους πείσω ότι δεν υπάρχει επικάλυψη. Ε, λέτε ότι πρέπει να υπάρξει έτσι και ένα, ένας φορέας ευρωπαίος, ευρωπαϊκός. Ε, γιατί ας πούμε η ISB ε, κυριαρχείται τους Αμερικανούς. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν ένα αντίβαρο ευρωπαϊκό, λέτε εσείς. Αλλά πώς μπορώ να πείσω τους πολίτες ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο. Ο κ. Κλίντς. Κατά την άποψή μου είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς την ΕΦΡΑΓ. Γιατί τότε δεχόμαστε αυτό που μας ε, υποδεικνύει ο, Διεθνής, Οργανισμός Διεθνής, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Οτιδήποτε πει, οποτεδήποτε ας πούμε πει να ένα πρότυπο, χωρίς καμία προσαρμογή, χωρίς κανένα προβληματισμό, χωρίς να το προσαρμόσουμε στην ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα, το καταπίνουμε. Άρα τότε ουσιαστικά εξαρτώμαστε από ένα συμβούλιο που στο παρελθόν είχε επισύρει πολλές επικρίσεις. Και προς το παρόν δεν βλέπω καμία δυνατότητα να προχωρήσουμε ε, χωρίς την ΕΦΡΑΓ. Η ΕΦΡΑΓ είναι η ευρωπαϊκή προσέγγιση, η ευρωπαϊκή λύση για να επηρεάσουμε άμεσα τα πρότυπα όπως προτείνονται από τον Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Λονδίνου. Αν δεν το είχαμε, αν δεν είχαμε την ΕΦΡΑΓ, τι θα λέγαμε, το δεχόμαστε το πρότυπο ή το απορρίπτουμε. Δεν είναι σωστή αυτή η λύση. Στο παρελθόν, σωστό, σωστά είπατε ότι τα περισσότερα πρότυπα που προτάθηκαν από το Λονδίνο τα δέχτηκε, τα, επικύρωσε η ΕΦΡΑ και τα σωμάτωσε. Αλλά τώρα βλέπουμε όλο και μεγαλύτερη βούληση να υπερασπιστεί πιο άμεσα, πιο ανοιχτά την ευρωπαϊκή, τις ευρωπαϊκές θέσεις όταν χρειάζεται. Και στο μέλλον θα δούμε και διαφορές ανάμεσα στις προ, προτάσεις του οργανισμού του Λονδίνου και την τελική θέση, το τελικό πρότυπο που θα εφαρμοστεί στην Ευρώπη. Και αυτό θα γίνει χάρη στη δουλειά της ΕΦΡΑΓ. Προς το παρόν λοιπόν δεν βλέπω καμία δυνατότητα να καταργήσουμε την ΕΦΡΑΓ. Κατά την άποψή μου η έκθεση Μάισταντ δεν λέει κάτι τέτοιο. Δεν λέει ότι υπάρχει οργανισμός του Λονδίνου, γιατί λοιπόν να μην καταργήσουμε τους άλλους οργανισμούς. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα της έκθεσης Μαϊστά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κλίντς. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη ζήτηση για τις πολλές ερωτήσεις που έκαναν και σένα για τις απαντήσεις. Πριν ε, περάσουμε στην κεκλεισμένη των θυρών ε, πλευρά της συνεδρίασής μα. Ήθελα να χαιρετήσω τον κύριο Όλη Σμιτ που μόλι ήρθε εδώ. Όλοι καλώς ήρθες. Ωραία. Οπότε τώρα παρακαλώ όλοι όσοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν κατά την ε, κεκλεισμένη των θυρών συνεδρίαση να ε, αποχωρήσουν. Είναι λοιπόν μόνο οι βουλευτές, η γραμματεία της Επιτροπής και οι συνεργάτες των ε, βουλευτών.